Dear Φίλοι, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε. Ε, δεν έχω τα χαρτιά μου εδώ. Για δώστε μου. Συγγνώμη. Συγγνώμη, λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως. Έχουμε διήμερη συνεδρίαση βεβαίως. Αν δεν υπάρχουν όλα σχόλια η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Δεν βλέπω δεν υπάρχουν σχόλια. Δεν έχω καμία ανακοίνωση. Εκτός από μία. Θυμάμαι και θα πρέπει και εσείς να θυμάστε ε, την ακρόαση της 21ης ε, ε, Φεβρουαρίου για την οδηγία για το αέριο και τις σχετικές τροπολογίες. Εντάξει. Γιατί προετοιμάζουμε την ακρόαση με τους συντονιστές 21 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, έχετε έναν μήνα. Έγκριση των πρακτικών, μάλιστα. 27 και 28 Νοεμβρίου, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της ε, συνεδρίασης, τα πρακτικά εγκρίνονται. Περνάμε τώρα στο σημείο 4. Δημόσια ακρόαση για το μέλλον της πολιτικής ε, της αμυντικής βιομηχανίας. Όπως ξέρετε είναι μια νέα ιδέα να υπογραμμίσω και πάλι ότι οι συνάδελφοί μας ε, από την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ την υποεπιτροπή αυτή της Επιτροπής Εξωτερικών ξεκίνησαν μία συζήτηση. Βεβαίως η πολιτική αυτή είναι ευθύνη της Επιτροπής Εξωτερικών αλλά η βιομηχανική πτυχή του θέματος είναι δική μας ε, ευθύνη προφανώς Οπότε είμαστε υπεύθυνοι για την προετοιμασία όλων των δράσεων που έχουν να κάνουν με την βιομηχανία. Πολύ σημαντικό αυτό και σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Βεβαίως έχουμε εδώ και τον κύριο εισηγητή ε, και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ε, τώρα όμως να πω ότι έχουμε και τους ομιλητές μας διακεκριμένος και θα συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους μας ειδικού. Εργάζονται οι δύο επιτροπές ε, ε, επί της πρότασης της Κομισιόν. Πρόκειται για το πρώτο νομοθετικό αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Για το επόμενο ΠΔΠ η Κομισιόν θα υποβάλει μια νομοθετική πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα που θα συνοδεύεται από μια πρόταση για ένα πρόγραμμα έρευνας της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Και βέβαια έχουμε εδώ πέρα και το άρθρο 54 του κανονισμού με την Επιτροπή Προπολογισμού και βεβαίω ε, και σε συνεργασία με την ΣΕΝΤΕ. Γιατί εντάξει, ε, τη ΣΕΝΤΕ αφορά και θα ξοδεύσουμε και λεφτά. Οπότε να καλωσορίσω την κυρία Φρανσουάζ Γκοστέτ, που εισηγήτρια. Από την Επιτροπή Προπολογισμού έχουμε τον κύριο Κοζάλης Πόνς, είναι εδώ. Δεν τον βλέπω. Μάλλον θα έρθει μετά. Και... Και Ζιόν Πάσκο, εισηγητής της ΑΦΕΤ. Δεν τον βλέπω ακόμα. Έχουμε επίσης έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής των Περιφερειών, τον κύριο Τούλε. Ωραία, σας ευχαριστώ. Έχουμε δυόμιση ώρες στην διάθεσή μας για τη συζήτηση αυτή. Και αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω τους ειδικούς μας. Παρακαλώ να μην ε, μιλήσετε για πάνω από 10 λεπτά γιατί θέλουμε να γίνει μια συζήτηση. Καλύτερο είναι να προσθέσετε κάτι ε, μετά. Λοιπόν, πρώτος ε, ομιλητής ο κύριος Γιάννη Πία, γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Αεροδιαστημικών και Αμυντικών Βιομηχανιών της Ευρώπης. Όπως ξέρετε, βασιζόμαστε στις βιομηχανίες αυτές. Θα θέλαμε να δείξουμε κάποιες ιδέες. Από την άλλη, θέλουμε για να τους στηρίξουμε. Αγαπητέ φίλε, λοιπόν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ και τα μέλη τη Επιτροπή ε, Χαίρομαι που είμαι εδώ εκ μέρου τη βιομηχανία για να αναφερθώ στο σημαντικό θέμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματο Βιομηχανική Ανάπτυξη στην Άμυνα. Ξέρουμε ότι κατατέθηκαν οι προτάσει ε, τον πρισμήν Ιουνίου και το Συμβούλιο κατέληξε γενική προσέγγιση το Δεκέμβριο και τώρα το Κοινοβούλιο παρουσιάζει την, ε, προετοιμάζει την εκθεσή του. Εγώ δεν θα αναφερθώ στα διάφορα έγγραφα, αλλά θα προσπαθήσω να υπογραμμίσω διάφορες αρχές ε, που θεωρούνται πολύ σημαντικέ από τη δική μας σκοπιά της βιομηχανίας. Συγγνώμη, είναι και... Έχω και ένα θέμα με το λαιμό μου σήμερα για να σας πω τι κρύβεται πίσω από το όνομα ESD. Όπως γνωρίζετε είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της αμήνας και των στρατηγικής. προσωπούμε πάνω από 300 εταιρείε από το βορρά στο νότο, από την Ανατολή στη Δύση, σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε 24 εθνικές οργανώσεις που προέρχονται από 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε εθνικές ενώσεις από την Ορβηγία και την Τουρκία. Επιπρόσθετα έχουμε 15 πολυεθνικές εταιρείες που είναι άμεσα μέλη της ESD ό,τι αφορά τις εθνικές ενώσεις. Ε, φυσικά ε, οι περισσότερες είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, και έχουμε και 10 ενώσεις στο επίπεδο του Συμβουλίου. Προς ε, το παρόν έχουμε Σουηδία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ολλανδία, Αυστρία ε, στο Συμβουλίο. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. Εκπροσωπούμε την, Ευρώ, την ε, ευρύτερη ευρωπαϊκή βιομηχανία, τις μεγάλες, μεσές και μικρές εταιρείες και έχουμε μια ευρεία γεωγραφική κατανομή. Καταρχήν, λοιπόν, η βιομηχανία μας υποστηρίζεται, υποστηρίζει το Ταμείο για την Άμυνα. Έτσι, λοιπόν, υποστηρίζουμε το πρόγραμμα έρευνας για την άμυνα και το πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στην άμυνα. Γιατί? Καταρχήν, η βιομηχανία μας είναι ανταγωνιστική και αυτή είναι μια δηλώση κλειδί. Έχουμε πολύ καλά προϊόντα παγκοσμίω και ήμασταν στην ακμή της τεχνολογίας και είναι πλήρως ανταγωνιστικά ε, όμως ε, αυτή είναι η καρπή ε, κάποιων επενδύσεων που έγιναν στο παρελθόν. Ε, στο μέλλον ε, δεν υπάρχει τίποτα για να αναπτυχθεί ή για να, παραμείνει, να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, αν θέλετε. Έτσι λοιπόν, παρά τα χρήματα που δαπανούνται στην Ευρώπη, δεν έχουμε αποτελεσματική εσωτερική αγορά. Πρέπει να δούμε ποιε θα είναι οι τεχνολογίε επόμενη γενιά σε πολλού τομεί. Ήδη βλέπουμε κάποιε ελλείψει στι ευρωπαϊκέ ενόπλε δυνάμει. Η απάντηση λοιπόν στην κατάσταση αυτή ζητά νέα προγράμματα. Χωρίς νέα προγράμματα δεν ε, θα υπάρχει ανταγωνιστικότητα μακροπρόθεσμα δεν θα είναι δυνατό να μείνουμε ε, στην ε, κορφή της τεχνολογίας, ούτε θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις δεξιότητες ε, και την τεχνογνωσία μας. Και όταν χαθούν αυτές οι δεξιότητες θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις οικοδομήσουμε εκ νέου. Από τη σκοπιά αυτή δεν χρειάζεται λοιπόν να πω ότι και η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία χάνεται αν υπάρξει με τέτοια εξέλιξη. Τα νέα προγράμματα είναι ζωτικά όχι μόνο για τα κράτη-μέλη και για ολόκληρη την Ευρώπη και την βιομηχανία. Αλλά πολλές ε, από αυτές τις προκλήσεις ε, είναι πολύ ακριβές και ιδιαίτερα απαιτητικέ σε εθνικό επίπεδο και αυτό ισχύει ε, κυρίως για τα πιο πολύπλοκα αμυντικά συστήματα. Και καθώς κανένα κράτος μέλος ε, δεν μπορεί μόνο του να το χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα, πρέπει να συνεργαστούμε. Αλλά εδώ δεν ε, μιλάμε για ένα οικονομικό εμπόδιο. Πολλά θα κερδίσουμε από αυξημένη συνεργασία και θα έχουμε και χαμηλότερο κόστος επιχειρησιακό. Όλοι γνωρίζουμε λοιπόν ότι δεν ε, είναι εύκολη η συνεργασία στον τομέα της άμυνας, αλλά αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα, θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε το EDF, το EDRP και το EDP όλα μαζί μπορούν να κάνουν ε, τη διαφορά η χρηματοδότηση για την ε, έρευνα στον τομέα της άμυνας μπορεί να δημιουργήσει ε, τη συνορική συνεργασία μεταξύ κρατών, ε, να ενισχύσει τη συνεργασία για την τεχνολογική αριστεία και αυτά τα δύο συνδυασμένα βάσει της φύσης τους θα μας δώσουν μια στρατηγική αυτονομία. Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη είναι σημαντικές γιατί θα καλύψουν την κοιλάδα του θανάτου εδώ πάρα πολλά προϊόντα πέθαναν ε, στο παρελθόν λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης ή λόγω της έλλειψης εναρμόνισης των απαιτήσεων. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό υποστηρίζουμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανική Ανάπτυξη στην Άμυνα. Το EDP όμω πρέπει να είναι φιλόδοξο, θα πρέπει να είναι ε, μεγάλο σε μέγεθο. Και γι' αυτό εμεί συμφωνούμε με την πρόταση τη Κομισιόν ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να είναι 500 εκατομμύρια ευρώ για το 2019 και το 2020 και να έχει ε, μια φιλοδοξία για να φτάσουμε στο επίπεδο του ενό δισεκατομμυρίου του χρόνου. Αυτό θα κάνει τη διαφορά, όμω δεν θα μπορέσουμε να είμαστε κάτω από αυτό. Έτσι λοιπόν, αν εγκριθεί αυτός ο προϋπολογισμός, ε, θα ε, αυξήσει τις δαπάνες στην Ευρώπη για την άμυνα και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Όμως δεν έχει να κάνει με το πόσα χρήματα δαπανάμε, αλλά και με το πώς. Πρέπει να δαπανίσουμε πιο αποτελεσματικά ε, τα χρήματα είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την συνέπεια, συνέχεια μεταξύ του ADP και των άλλων προγραμμάτων σε επίπεδο κρατών μελών. Πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και για τα δύο σκέλη του Ταμείου Άμυνας θα πρέπει να σχεδιάσουμε από κοινού και τα δύο προγράμματα και θα πρέπει να συντονίζεται το σχέδιο των επενδύσεων με τα επενδυτικά των μελών και να τα συμπληρώνει με το σωστό μηχανισμό και τις ε, δομές η ευρωπαϊκή συνεργασία θα κάνει ένα τεράστιο βήμα προς τα μπρος. Επιπλέον, για να κάνουμε μια διαφορά. Δεν μιλάμε μόνο για το επίπεδο τη χρηματοδότηση και του σχεδιασμού, αλλά και πού φυσικά δαπανά κάποιο τα χρήματα. Θα πρέπει να δαπανίσουμε τα χρήματα στο να αναπτύξουμε ικανότητε που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, μια επιχειρησιακή διαφορά και τεχνολογική διαφορά. Θα πρέπει εδώ να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια διαδικασία που θα ε, βρίσκει ποιε είναι οι ανάγκε των κρατών μελών ω προ τι ικανότητε και θα πρέπει να εντοπίσουμε, να ταυτοποιήσουμε κάθε μία από αυτέ τι ανάγκε που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη συνεργασία. Επίση, ε, τα χρήματα θα πρέπει να πηγαίνουν σε ευρωπαϊκέ βιομηχανίε. Αυτό είναι σημαντικό για πολιτικού λόγου, για λόγου ασφάλεια και κατόπιν ε, ερχόμαστε ε, στο θέμα αυτό ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ε, εταιρεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι τεχνολογικέ ικανότητε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η τεχνογνωσία που χρηματοδοτείται από την Ένωση θα παραμείνει εντό τη Ένωση. Πώ θα το πετύχουμε αυτό. Αυτό συνεχίζεται στην νομοθετική διαδικασία και μπορεί να επανέλθουμε αργότερα στι ερωταπαντήσει. να πω και κάτι σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και τη συμπερίληψη. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι κάτι που θα πρέπει να ωφελήσει όλα τα μέρη της αλυσίδας ε, προμήθειας, ε, μικρές ε, και μεγαλύτερες εταιρείε. Όλοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ευκαιρία για πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Επίσης, η αποτελεσματικότητα του προγράμματος δεν μπορεί να διακυδευτεί. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε εξισορρόπηση εδώ. Θα πρέπει να διατηρηθεί η βιομηχανική ηγεσία, αλλά θα πρέπει να ε, έχει και όλη την ευθύνη αυτός που θα αναλάβει το συμβόλαιο για την ε, αλυσίδα εφοδιασμού. Ε, μόνο αν η αλυσίδα εφοδιασμού είναι ανταγωνιστική μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικότητα σε συνολικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι το EDP θα πρέπει αφενός να προωθήσει τη διασυνοριακή βιομηχανική συνεργασία και να διασφαλίσει ότι η τεχνολογική και βιομηχανική λογική διέπει το πρόγραμμα. Ε, εξίσου σημαντικό, οι κανόνε για τη χρηματοδότηση, όπω ξέρουν όλοι, δεν είναι εμπορική αγορά η άμυνα. Οι κυβερνήσει είναι οι μόνοι πελάτε των προϊόντων τη Άμυνα, και είναι αυτέ που θα αποφασίσουν για τι εξαγωγέ. Επομένω, μια εταιρεία που δρά ω οικονομικό φορέα δεν μπορεί να θέσει τα δικά τη χρήματα επιτόπου χωρί να έχει δέσμευση από τον πελάτη ότι θα αγοραστεί το προϊόν. Και για να το πω ξεκάθαρα, μπορεί να σκοτώσει μια εταιρεία αν θε να λάβει τέτοιου κινδύνου. Και αυτή είναι μια γνωστή ιδιαιτερότητα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στο προγράμματα ανάπτυξη και έρευνα στην άμυνα. για το EDP, Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για επιλέξιμο κόστος αφενός ε, και του πραγματικού συνολικού κόστους, ε, από την άλλη θα πρέπει να καλύπτεται από τα κράτη-μέλη. Η ιδιαιτερότητα της ε, αγοράς άμυνας ισχύει, ισχύει και για τις ε, εξαγωγές και για το EIPR. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σεβαστούμε την ευθύνη των κρατών μελών, να αναλαμβάνουν τις αποφάσεις για τις εξαγωγές. Τα EIPR θα πρέπει να παραμένουν τα δικαιώματα πνευματικής διοκτησίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται μόνο όταν έχει τελειώσει η κυριότητα ενός ε, project. Οι αποφάσεις για εξαγωγή ε, είναι κάτι που εναπόκειται μόνο στα κράτη-μέλη. Και για να λήξω με μια τελευταία διαφάνεια. Θα συνοψίσω ω εξή. Είναι ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή βιομηχανία βάσει των επενδύσεων του παρελθόντο. Ε, αν, ε, βάλουμε, αν ε, προσθέσουμε τι δαπάνε των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δεύτερη αγορά παγκοσμίω, όμω δεν έχει τη δυνατότητα να ξεκλειδώσει τη δυναμική τη για να παραμείνει παγκόσμιο παίκτη, γιατί τώρα δεν έχουμε κάτι για το μέλλον. Δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστική μα θέση και γι' αυτό υποστηρίζει η βιομηχανία το πρόγραμμα έρευνας, το πρόγραμμα ανάπτυξης στον τομέα της ε, άμυνας ε, ε, το EDP είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος από οικονομική και πολιτική σκοπιά. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας, για τα σχόλιά σας. Επόμενος ομιλητής, ο κ. Γιάκομπ Λαντόφσκι, Υφυπουργός Αμήνης Τεχικής Δημοκρατίας. Να προσθέσω κάτι. Στον πρώτο γύρο της ακροάσεως θα ακούσουμε εκπροσώπους της βιομηχανίας και εκπροσώπους των κρατών μελών. Απόψεις κρατών μελών και βιομηχανίας. Στο δεύτερο τμήμα των συζητήσεων της ακροάσεως πάμε προς προγράμματα βιομηχανικής αναπτύξεως στον αμυντικό τομέα κάτι στο, για το οποίο θα μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά αμυντικά ερευνητικά προγράμματα. Θα είναι νομοθετική πρόταση που αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το επόμενο. Στο δεύτερο τμήμα λοιπόν θα συζητήσουμε το όλο ζήτημα με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών επιστημονικών κύκλων, ερευνητές επιστήμονες. Το δεύτερο τμήμα θα αφορά περισσότερο την ε, έρευνα, ανάπτυξη και ενοτομία του μυντικού τομέα. Τώρα ακούμε την άποψη της βιομηχανίας και των κρατών μελών. Η τσεχική δημοκρατία λοιπόν. Ο Υφυπουργό Άμυνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για το λόγο, κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Μεγάλη τιμή για μένα που μιλώ στην Επιτροπή. Η ομιλία μου θα εκφράσει τις απόψεις για τις τρέχους εξελίξεις και μελλοντικές προοπτικές όπως τα βλέπει η Τσεχία. Είναι ένα από τα μικρότερα κράτη-μέλη. Θα ξεκινήσω από το συνέστημα που έχω διαμορφώσει στι Βρυξέλλες. Έφτασα νωρίς το πρωί και αισθάνομαι ότι υπάρχουν προσδοκίες όσον αφορά το νομοθέτημα. Είναι σχεδόν απτές οι προσδοκίες. Δεν θα κρυθούμε μόνο από τις επιτυχίες μας και από τα χρήματα που θα δαπανίσουμε αλλά θα κρυθούμε εν συγκρίση με την πλούσια παράδοση της αμυντικής, ε, του αμυντικού τομέα στην Ευρώπη που έχει ξεκινήσει προσπάθεια στην δεκαετία του 50. Πολλά έχουν ανάξει δεκαετία του 50. Να λάβουμε υπόψη τις πολύ διαφορετικές απειλές σημερινές συγκρίσει με τη δεκαετία του 50 και πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τις αμυντικές δαπάνες που ανταποκρίνονται τις ε, απειλές. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Και μπορούμε να δούμε ε, από οπτική γωνία κάθε χώρα γιατί ακολουθούμε αυτή την προσέγγιση. Τώρα έχουμε κοινή στρατηγική, μια γενική ε, ευρωπαϊκή στρατηγική και πρέπει να βρούμε τρόπο να προωθήσουμε τη στρατηγική την ευρωπαϊκή στον κόσμο. Για να είμαστε επιτυχείς πρέπει να βρούμε και τον τρόπο με τον οποίο συνδέσουμε τη στρατηγική με το παρόν αμυντικό πλαίσιο της Ευρώπης αποτελείται κυρίως από το ΝΑΤΟ. Όποτε μιλάω για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, αναφέρομαι σε δυστυχία. στοιχεία. Διότι μιλάμε για συμπληρωματικότητα και αξιοπιστία. Βασικές στοιχεία. Συμπληρωματικότητα μπορεί να επιληθεί αν υπάρχει σωστός επιμερισμός των ρόλων και αξιοπιστία που εξαρτάται από το αποσά που διαθέτουμε για τις αμυντικές δαπάνες. Πρώτο αναγκαίο βήμα. Να εξετάσουμε τα αντιμετωπιζόμενα προβλήματα στα πλαίσια της στρατηγικής μας. Έχουμε αυτή την διαμόρφωση της νέας στρατηγικής για να έχουμε έρευνα και ανάπτυξη και παραγωγή που ταιριάζει με τους στόχους μας. Θέλουμε να έχουμε την πιο ποιοτική τεχνολογία της δυνάμεις παρά το κατακαιρματισμένο κεφάλαιο και παραγωγή του αμυντικού τομέα στην Ευρώπη. Το ανέφερε προλαλή σα. Θέλουμε να ενοποιήσουμε την αμυντική βιομηχανία για να είμαστε αποδοτικότεροι οικονομικά. Πρέπει να δούμε όμω ότι ξεκάθαρα και ποια είναι οι δυνατότητε των αμυντικών μα, των όπλων μα δυνάμεων. Γιατί χρειάζονται οι ενόπλε δυνάμει. Η πρωτοβουλία τη ΠΕΣΚΟ είναι μια καλή αφετηρία. Είναι η γίδα για όλε τι ε, εξελισσόμενε πρωτοβουλίε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τους πόρους, να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες διαλειτουργικές τεχνολογίες. Χρειάζεται καλύτερη συμβατότητα από ό,τι κατά παρελθόν. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι πόρο απέχουμε από το βασικό στόχο. Να έχουμε ένα σαφή, σαφές όραμα όσον αφορά την ενοποιημένη αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε έναν πελάτη, ενίο πελάτη και έναν χρήστη. Πρέπει να εξετάσουμε διεξοδικά αν θέλουμε η βιομηχανία μας να αναπτυχθεί μόνο και μόνο για να ισχυροποιηθεί. Ή αν θέλουμε μια πληρέστερη αμυντική αγορά επίσης. Είναι ακρογωνίως λήθος αυτή η απόφαση. Πάνω σε αυτό το λίθο θα στηριχθούν τα επόμενα βήματα. Ήδη υπάρχει εξέλιξη. Όλοι κατανοούμε ότι χρειάζεται βήμα-βήμα να οικοδομήσουμε μια πληρεστερη αμυντικη αγορα επισης ειναι ακρογωνιως λιθος αυτη η αποφαση πανω σε αυτο το λιθο θα στηριχθουν δομή Χρειάζεται συμμετοχή των κατών μελών. Χρειαζόμαστε μέτρα κατάλληλα να συμμετέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μέσω μέτρων που ήδη έχουν προταθεί για το EDDIP. Εμείς υποστηρίζουμε ένθερμα και την ΠΕΣΚΟ και την EDIP. Οι σχετικές πρωτοβουλίες στηρίζουν προγράμματα ΠΕΣΚΟ και έχουμε πάνω από 12 προγράμματα έτοιμα. Η αμυντική μας βιομηχανία ισχυροποιείται και σε μέγεθος και σε αριθμό συμμετεχουσών εταιριών και κέρδη. Είμαστε εξαγω... στεφόμαστε προς τις εξαγωγές. Οι εξαγωγές μας έχουν τριπλασιαστεί περίπου την τελευταία πενταετία. Η διεθνή συνεργασία είναι πολύ σημαντική για μας και πρέπει να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στους κύκλους εφοδιασμού και να δημιουργήσουμε και νέους χώρους. Χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Είναι κλειδί για βέλτιστο, ε, βέλτιστη ασφάλεια εφοδιασμού για τι αναπλέ δυνάμεις. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα. Χρειάζεται αμοιβαία συνεργασία λόγω αλληλεξάρτηση. Πάνω από 90% ανοίξει τον ιδιωτικό τομέα βιομηχανία μα. Κατανοούμε άριστα ότι υπέθετηθούν σωστέ ισορροπημένε προσεγγίσει που θα ανταποκρίνουν τι των ενόπλων μα δυνάμεων και ταυτόχρονα να διαπνέονται από επιχειρηματικό πνεύμα. Πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο ε, νομοθετικό πλαίσιο που θα δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδοσιακά είχαμε βασιστεί στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Πρέπει να είναι διάφοροι ορισμοί που θα εφαρμόζονται σωστά. Ε, ο ορισμό των μικρομεσαίων είναι πάνω ε, μάλλον μέχρι 250 εργαζομένου. Παρά τι προσπάθειε που κάνουμε, οι εταιρείε δεν μπορούν να γίγονται όμως όπως η Airbus ή η British Aerospace ή η KMW. Άρα έχουμε νέα κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων που θα στηρίζεται μέσω του EDDIP ε, όπως και οι μικρομεσαίες. Έπρεπε λοιπόν να έχουμε φύστατη για να ακολουθήσουμε για να προωθήσουμε τη βιομηχανία και να ανταποκριθούμε σαν ανάγκε των όπλων δυνάμεων. Γι' αυτό υιοθετήσαμε στατηγική για υποστήριξη εφοδιασμού στην Τσεχία πάνω στις ίδιες αρχές που προανέφερα και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι η αμυντική βιομηχανία είναι στατηγικό τομέα. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το ίδιο όπως άλλοι τομεί. Είναι ένα στο τμήμα αμυντικών οικοσυστημάτων. Άρα χρειάζεται μια συγκεκριμένη πολιτική. Πρέπει να εξετάσουμε την πολιτική, να διαμορφώσουμε σωστά, να μην επηρεάσουμε τις επιχειρήσεις του τομέα, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις ανάγκες των βασικών χρηστών. Και πρέπει να καθορίζονται αυτές οι ανάγκες στα συμφέροντα των πρωταρχικών χρηστών. Είμαστε κοντά στους στόχους. Η τσεχική βιομηχανία μέσω των πρωτοβουλειών που έχει εφαρμόσει έχει προβεί σωστή αξιολόγηση, έχει αξιολογηθεί από τους αιτητικούς Είμαστε σε διάλογο με τις χώρες εταίρους, με τη Σλοβακία, την Ιταλία, τη Γερμανία, Ισπανία και με την Αυστρία στι προσπάθειε που καταβάλουμε. Και συζητούμε το πώς θα έχουμε το πιο δίκαιο και διαφανές σύστημα για τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Και θα πρέπει να έρχομαι σε επαφή με τους αρμοδίους της Γενικής Διευθύνσεω Γκρο. Ενδιαφερόμεθα πολύ να ακούσουμε τις απόψεις του Ευρωκοινοβουλίου. Τις απόψεις σας κυρίες και κύριοι. Θα σταματήσω εδώ την ομιλία μου και θα είμαι έτοιμος να ακούσω τυχόν ερωτήσεις που θα με επευθυνθούν. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you for your speech and your σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Αν ε, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω την συζήτηση, αγαπητοί φίλοι, με την κυρία Γκροστέτ. Φρανσουάζ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Γράμματος ε, τις πολιτικές για την αμυντική βιομηχανία. Είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση Άκουσα τι είπε ο Γενικός Γραμματέας ε, της Ένωσης, ASD, Μα είπε ότι τα επιχειρήσει, προσπαθώντα φυσικά ταυτόχρονα να εξεύρουμε και νέε συνεργασίε με άλλου ε, ευρωπαίου εταίρου. Μίλησαμε για τι μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει, την διαρροή τη τεχνογνωσία μα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ερώτηση λοιπόν που θέτω εγώ, καθώ μιλήσαμε για ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, Πόμενα και των ξένων επενδύσεων. Μιλήσαμε για την ευρωπαϊκή επιχείρηση, για τον ορισμό τη ευρωπαϊκή επιχείρηση. Αυτό μάλιστα ήταν και αντικειμένο συζήτηση. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Μάλλον δεν έχουμε κανέναν από την ε, Επιτροπή Προπολογισμού. Είχε γίνει μια γνωμοδότηση βάση του άρθρου 54, το ίδιο ισχύει και για τη ΣΕΝΤΕ. Έχουμε όμως ε, κάποιον εκπρόσωπο από τη ΣΕΝΤΕ, δεν έχουμε και τον εισηγητή, αλλά αν θέλετε να πάρετε το λόγο τώρα εκ μέρου τη ΕΝΤΕ, όχι, αργότερα. Επομένω, α πάμε στι πολιτικέ ομάδε. Κύριο Πάχη, μέρου ε, των Σοσιαλιστών. Και σε ποιο βαθμό μπορεί η ιδιοκτησία αυτή ε, των εταιριών που βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορεί να περιγραφεί. Ε, τι θα πούμε, ότι θα πρέπει να έχουν Ευρωπαίους ιδιοκτήτες και πιο... δεν ξοδεύουν αρκετά στις ενόπλες δυνάμεις. Και φοβάμαι ελαφρώ ότι οι βουλευτές εδώ θα θεωρήσουν αυτό το πρόγραμμα ως υποκατάστατο για τις εθνικές τους δαπάνες. Η ερωτήση λοιπόν που θα έφτα εγώ είναι το πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπουτικόφερ, εξ των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελάτη σε μια μπειραρία που έπινε όλη η μέρα που το κερνούσε τον μπαρ και το ζητούσε και μπύρα περισσότερη και άλλα ποτά. Αυτή για τις προμήθειες ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο το 2009 και δεν εφαρμόζονται οι κανόνες. Ακούγοντάς σας, θεωρητική λογική για την αγορά αυτό το σκοπό έχει η οδηγία για τις ε, κρατικές προμήθειες και αντί να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση, εξοικονομώντας 25 μέχρι 100 δις το χρόνο για τους φορολογούμενους. Και εδώ απηχώ αυτά που είπε ο κύριος Φόξ. Πρέπει να εκπροσωπούν. Δεν είναι λύση. Ξοδεύουν πολλά χρήματα, αλλά δεν αξίζουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών, τα χρήματα που δίνουμε. Μέσω συγχωνεύσεων και κεντρικής διαχείρισης μπορούμε να πετύχουμε ανταγωνιστικότητα. Μπορούμε να ακολουθήσουμε βιομηχανικές προσεγγίσεις, εμπορικές, αντί να ρίχνουμε χρήματα. Και ερώτησή μου. Στο Κοινοβούλιο έχουμε τοποθετηθεί όσον αφορά κατηγορίες όπλων, όπως όπλα μαζικής καταστροφής, απεμπλουτισμένο ουράνιο, ε, απάνθρωπα όπλα κλπ. Θα θέλαμε να συνδέσουμε τα χρήματα που δαπανούμε για την άμυνα με σαφή θέση. Αυτή η θέση ποια είναι. Ότι δεν θα υπονομεύουμε τις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα. Και δεν θέλουμε να εξοδεύονται χρήματα για όπλα και μη πανδρομένα οχήματα πριν να έχουμε το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Συμφωνείτε με αυτά. Προς τον κύριο Υφυπουργό. Είπατε τον ακρογωνίο λίθο, την απόφαση που είναι ακρογωνίος λίθος της προσέγγισής σας. Θα συνεχίσουμε με κατακαιρματισμένους πελάτες και αγορά ή θα κινηθούμε προς μια ολοκληρωμένη αγορά. Εγώ καταρχάς θα υποστήριζα Πρέπει να δούμε τι βοηθά να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Τι θεωρείτε ότι μας βοηθά να πετύχουμε το στόχο. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή την πτυχή. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να εντοπίσουμε τα κατάλληλα μέτρα που θα μας οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι θα ξεπεράσουμε τη σπατάλη χρημάτων σε... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω τσεχικά. Και προς όφελος και του κυρίου Φιπουργού να ακούσει τη μητρική του γλώσσα πιστεύω ότι βασική και προδιαγραφές. Εγώ έχω ασχοληθεί με την παραγωγή γυαλιού και πριν από 100 χρόνια στον τομέα ε, του γυαλιού είχαμε κοινά πρότυπα, τσεχικά πρότυπα, γερμανικά πρότυπα τα οποία είχαν διαδοθεί και χρησιμοποιήθηκαν από άλλες χώρες. Στον αμυντικό τομέα δεν έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία ενός αναπτυξιακού κέντρου για την κατασκευή κινητήρων. Και πώς θα προστατεύσουμε το σχεδιασμό και τα πνευματικά δικαιώματα αν υπάρχει τεχνολογική εξέλιξη, ένας κινητήρας, ένα αεροσκάφος και έχει κάποιο ανταλλακτικό αμερικανικό το προϊόν, δεν εξάγεται το προϊόν σε ξένες αγορές. Αυτό κάνει οι Αμερικανοί. Τρίτον, η βασική τα υλικά χρειάζεται συντονισμός αυτής της βασικής έρευνας Παραδείγματο χάρη ξεκινάμε από τα θεθωρακισμένα οχήματα, στα όπλα ή καθευτή Αποτελείται από τα πορίσματα της βασικής έρευνας Πάμε στον τεχνικό σχεδιασμό, πάμε στον εξοπλισμό και τα μηχανήματα, hardware, και μετά έχουμε το λογισμικό, software. Έχουμε τρεις ξεχωριστούς τομείς. Πρέπει να επενδύσουμε συντονισμένα και στους τρεις τομείς. Ε, οι δαπάνες γίνονται για παράλληλες έρευνες. Έχουμε πετύχει στον τομέα στην προσέγγιση αυτή στην Τσεχία στην αεροναυπηγική, στην αεροπορική βιομηχανία δεν είναι απλά τα πράγματα. Παράγουμε πόρτες για τα Airbus, παραδείγματο χάρη. Όσον αφορά όμω το λογισμικό, εισάγουμε λογισμικό από άλλε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Πρέπει να δούμε λοιπόν προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Ο συνάδελφος ήδη είπε ότι τα χρήματα που διαθέτουμε θα πρέπει αντιμετωπίσαμε τη ΣΥΠΑ, ότι δεν μπορούσαμε να εξάγουμε αυτό που θέλαμε να εξάγουμε. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε αυτά τα λάθη και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκου, που είναι συντάκτης της γνωμοδότησης εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο θα ψηφίσουμε στην ΑΦΕΤ ε, και προετοίμαζα τον κατάλογο όταν ε, έμαθα ότι περιμένατε <laughs> μια γνωμοδότηση από τον ε, συντάκτη της γνωμοδότησης. Όπως γνωρίζετε, είχαμε 365 τροπολογίες, ε, προετοιμάσαμε 13 συμβιβαστικές που καλύπτουν την πλειοψηφία των τροπολογιών που κατατέθηκαν. Η φιλοσοφία μας ήταν να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία, όχι να σκοτώσουμε την πρωτοβουλία. Έπρεπε λοιπόν ε, να βρούμε μια εξισορρόπηση, μια ισορροπία αφενός του να διατηρήσουμε τη στρατηγική γραμμή, ότι πρέπει να υποστηριχτεί η πρωτοβουλία, αλλά ταυτόχρονα δεν θα έπρεπε να κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, δηλαδή να προσθέσουμε διάφορες μικρές τροπολογίες εδώ και εκεί. Έτσι λοιπόν έπρεπε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο. Υπήρχαν τροπολογίες που προσπαθούσαν ε, να εισαγάγουν κανονισμούς, κανόνες σε τομείς που δεν είναι αντικείμενο αυτή της πρωτοβουλίας. Πρέπει να το σχάρει τις εξαγωγές όπλων. Είναι ρυθμισμένες, υπάρχει ένας σχετικός κανονισμός. Έτσι λοιπόν δεν νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πίσω πόρτα για να επηρεάσουμε τους εφιστάμενους κανονισμούς για άλλους τομείς. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο οποίο εξακολουθούμε να προσπαθούμε να βρούμε λύση και νομίζω γνωρίζετε ότι μπορεί να έχουμε αύριο μια καλή λύση. Πέραν αυτών είχαμε συζητήσεις με τους και Ξέρουμε ποια είναι η στάση τους, έχουμε διαβουλευτεί μαζί τους και ανυπομονούμε για την ευρωιανή ψηφοφορία στις 11. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ο κύριος Γκάιερ από την Επιτροπή Συνταγματικών ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, είχαμε κάποια μείωση το 2012-2013, όμως τώρα βλέπουμε νέα αύξηση και γίνεται μια επένδυση στις ε, δαπάνες, στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Πώς σχετίζεται αυτό αυτή με την Ευρώπη. Αν επιβιώσεις ε, στους απλούς πολιτές ε, υπάρχει ε, και ισχυρή ευρωπαϊκή φιλοδοξία. Θα πρέπει να οικοδομηθεί η ευρωπαϊκή ικανότητα θα θέλουν να οικοδομήσουν τις δικές τους αμυντικές πολιτικές και τις ε, τεχνολογικές και βιομηχανικές βάσεις και ζητούν και για μεταβίβαση της τεχνολογίας. Αν τους βοηθήσετε να ε, δημιουργήσουν τις δικές τους αμυντικές βιομηχανίες είστε ευπρόσδεκτοι. Και υπάρχει και το θέμα τη μεταβίβαση τεχνολογία. Αν λοιπόν η στρατηγική επιβίωση βασίζεται σε εξαγωγέ, πώ θα το κάνετε αυτό όταν οι χώρε αυτέ ε, στι οποίε εξάγεται θα γίνουν οι μελλοντικοί ανταγωνιστέ σα, θα πρέπει να δείτε τι συμβαίνει και μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσετε σοβαρά στην έρευνα για να μείνετε στην κορφή τη αλυσίδα αξία. αν δούμε τις επιδόσεις της Ευρώπης, ε, θα δούμε ότι δεν είναι καλές. Αυτή είναι η λυπηρή απάντηση. Δεν έχουμε επενδύσει στην έρευνα και στην ε, ανάπτυξη. Θα δείτε ότι τα ευρωπαϊκά επίπεδα της ε, ε, χρηματοδότηση στην άμυνα είναι πολύ κατώτερα από άλλες περιοχές παγκοσμίω και σε ό,τι αφορά τον κατοικερματισμό της αγοράς. Καταρχήν συμφωνώ ότι δεν είναι λειτουργική αγορά και η οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες προσπάθησε να την κάνει να λειτουργεί καλύτερα. Και από την πλευρά της βιομηχανίας πιστεύουμε ότι αυτή η οδηγία ήταν μια καλή οδηγία. Παρ' όλα αυτά η εφαρμογή της δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο έπρεπε. Έτσι λοιπόν ε, συνεχίζουμε να πιέζουμε για πιο ε, ορθή, για πιο αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας. Όμως ε, θα πρέπει ε, η αλλαγή στη συμπεριφορά να αλλάξει από τα κράτη-μέλη. Δεν εξαρτάται από τη βιομηχανία. Δεν είναι αυτή η υπεύθυνη ε, για το να πουλήσει, παραδείγματος χάρη να έχει περισσότερα μοντέλα ελικόπτερο από ότι οι πελάτες που έχει για τα ελικόπτερα. Ουσιαστικά ο πελάτης καθορίζει και η βιομηχανία παράγει. Θα πρέπει λοιπόν από τους πελάτες να γίνει αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά και ακριβώ εδώ έρχεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μηχανικής Ανάπτυξη στην άμυνα. Αν έχουμε μια κατακαιρματισμένη αγορά, είμαστε ανταγωνιστικοί, ναι, αλλά επίση είπα τι σημαίνει το να είσαι ανταγωνιστικό, ότι μπορούμε ε, να προμηθεύουμε τι ικανότητε που ζητούνται από τι ευρωπαϊκέ ενόπλε δυνάμει σήμερα. Όμω αυτό βασίζεται σε επενδύσει που έγιναν στο παρελθόν. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι καινούριο στον ε, εγώ στην προετοιμασία, δηλαδή στο μέλλον δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί αν δεν υπάρχει νέο πρόγραμμα για να αναπτύξουμε την επόμενη γενιά τεχνολογιών. Επιπλέον, χάνουμε δεξιότητες στις εταιρείε αν ε, δεν υπάρχουν ε, τέτοια προγράμματα και δεν θα μείνουμε στο επίπεδο που είμαστε. Θέλουμε να αποφύγουμε ε, ουσιαστικά την ύφεση γιατί θα χάσουμε τα προσόντα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, Πιστεύουμε ότι το 1 δισεκατομμύριο στο επόμενο πρόγραμμα που έχει ζητηθεί ως κίνητρο για την αυξημένη συνεργασία δεν είναι υπερβολικό σκεφτείτε ότι δαπανούμε και 190 δισεκατομμύρια συνολικά. Δεν ζητάμε χρήματα λοιπόν για να διευρύνουμε την βιομηχανία. Απλώς ε, θα θέλαμε να προμηθεύουμε τα προϊόντα και τις ικανότητες που ζητούνται από τις ένοπλες δυνάμεις ούτε καν να εξαρτώμαστε από τις εξαγωγές. Βέβαια αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Έτσι λοιπόν καταρχήν πιστεύω ότι ε, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι ένα εργαλείο για να δώσει κίνητρα για τη συνεργασία. Η συνεργασία θα ήταν μια καλύτερη συμπεριφορά ε, ως προς την αγορά, περισσότερη αξία για τα χρήματα, περισσότερες ικανότητες για ε, το ίδιο επίπεδο των ποσών που δαπανώνται. Τώρα για να έρθω στις ερωτήσεις, τι γίνεται με την επιλεξιμότητα καταρχήν θα ε, έλεγα ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δράσει θα πρέπει να γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί έλεγχοι από τρίτε χώρε ε, επί τη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη δράση ή προκαλείται μέσα από τη, ή παράγεται μέσα από τη δράση, αν έχουμε μια οντότητα η προκαλειται μεσα απο παραγεται μεσα απο τη ανήκει σε τρίτη χώρα και η προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών ε, θα πρέπει επίσης να επιτυγχάνεται. Όλα αυτά θα πρέπει να συσταθούν για να διασφαλίσουμε μια σειρά. Τα δικαιώματα πνευματική διοκτησίας πρέπει να μείνουν εντό τη Ένωση. και αυτή η διαβεβαίωση θα πρέπει να έρθει και από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ο μηχανισμό που πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από πού θα έρχονταν τα χρήματα. Θα έλεγα ότι από τη βιομηχανία δεν είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να αποφασίσουμε από πού θα έρθουν τα χρήματα. Για μας είναι πιο σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι αν θέλετε να δώσετε κίνητρα ε, για την ανάπτυξη των ε, συνεργατικών ε, project, θα πρέπει να μιλάμε για ένα επαρκές ποσό για να κάνουμε τη διαφορά και ε, είχαμε ε, προσπαθήσει σε μια πρώτερη ομάδα που υποστηρίζεται και από την Κομισιόν ε, να προσδιορίσουμε ποια είναι αυτά τα επίπεδα και το 1 δισεκατομμύριο για ένα πρόγραμμα follow-on 250 εκατομμύρια εδώ πριν το χάρη είναι αρκετά για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία όμως αυτά θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά με τις επενδύσεις των κρατών μελών δεν θα έχουμε μείωση δηλαδή σε επίπεδο κράτους μέλους γιατί διαφορετικά θα χάναμε σε σχέση με το θέμα του αν είναι εμπορική αγορά. Μπορούμε να μιλάμε πολύ για τις ε, συνθήκες στην αγορά, όμως εδώ δεν έχουμε κάτι που να μοιάζει με εμπορική αγορά, αφενός. Μόνο η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι αγοράζει τα προϊόντα σου και δεύτερον είναι αυτοί που θα πούν αν ε, μπορείς ή όχι να εξάγεις. Και αν πιστεύεις ότι θα έχεις έγκριση τη κυβέρνηση για εξαγωγή, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να πουλήσει ε, ε, παντού σε όλο τον κόσμο ή ακόμη και στις χώρες που θα έχει εγκρίνει η κυβέρνηση. Γιατί, και αυτό είναι ενδιαφέρον, αν δεις που εξάγουν οι διάφορες χώρες, θα δεις ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο μοντέλο ε, για το ποιος είναι οι σχέσεις μεταξύ των χωρών. Έτσι λοιπόν οι συνθήκες της αγοράς δεν υπερισχύουν, δεν επικρατούν ε, στην αμυντική βιομηχανία. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να πληρώσουν οι χώρε για το επίπεδο αμύνας που θέλουν. Επανερχόμαστε λοιπόν στο θεμελιώδες ερώτημα. Θέλετε ευρωπαϊκές ενόπλες δυνάμεις ε, που να είναι καλά εξοπλισμένες, θέλετε αυτός ο εξοπλισμός να είναι ευρωπαϊκός ή θέλετε να εξαρτάστε από τους ε, Αμερικανού, του Ρώσους κτλ. Yeah. Uh, thank you very much. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να δημιουργήσουμε και δουλειές βέβαια στην Ήπειρό μας. Αλλά είναι ένα πολύ στη διάθεσή σας και για άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Θα παραμείνετε εδώ και στο δεύτερο τμήμα των συζητήσεων ίσως μπορείτε να λάβετε το λόγο. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Επιστημονικά ιδρύματα εκπροσώπη αυτών. από την ομάδα για την έρευνα, μάλλον για τις πληροφορίες, για την ειρήνη και την ασφάλεια. Παρακαλώ, όχι παραπάνω από 10 λεπτά, κύριε Μάρο. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε για να συμμετάσχω στον όλο προβληματισμό που εμπνέεται αυτό το πρόγραμμα και θα μιλήσω με ανεξαρτησία και ειλικρίνεια, τακτοποιώντας και στρέφοντα ιδέες μου γύρω από τρει παρατηρήσει βασικά. Η πρώτη είναι ότι όπω βλέπω εγώ τα πράγματα, ε, αυτή η προσέγγιση που ακολουθούμε είναι η καλύτερη απάντηση στην Ευρωπαϊκή Αμήνα εδώ και καιρό. Και δεύτερο, νομικά δεν έχω αμφιβολία ότι το πρόγραμμα αυτό συνάδει με τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Τρίτον, θέλω να πω ότι το μονοπάτι που επιλέξατε θα είναι μακρόν με πολλά εμπόδια και θα πρέπει να είστε υπομονετικοί και να επαγρυπνείτε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την πρώτη παρατήρηση. Το EDIDP είναι ό,τι καλύτερο για την Ευρωπαϊκή Άμυνα ε, και αυτό για δύο λόγους. Ε, το πρώτο είναι ότι αυτό το πρόγραμμα είναι στα χέρια των Ευρωπαϊκών Αρχών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, στα χέρια του Κοινοβουλίου που είναι τα μόνα όργανα που μπορούν να εκφράσουν το όραμά του που βασίζεται στα συμφέροντα τα ευρωπαϊκά που είναι κάτι παραπάνω από τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή των συμφερόντων των κρατών μελών αυτό διότι αυτέ οι αρχέ λαμβάνουν τι αποφάσει του με πλειοψηφία. Λοιπόν, η δημιουργία της ΠΕΣΚΟ τέλο 2017 κατέδειξε ότι με το άθροισμα δύο στοιχείων τα κράτη-μέλη δεν είναι πάντα σοβαρά όσον αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα ε, υποκρίνονται ότι είναι σοβαρά. Η μόνη χρησιμότητα της όλης ιστορίας είτε να δείξουν μια εικόνα στο εξωτερικό ότι είναι ενωμένοι οι Ευρωπαίοι, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα, και να πιστέψουν οι Ευρωπαίοι πολίτε ότι οι ηγέτε ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή Άμυνα συλλογικά, ενώ αυτό δεν αληθεύει. Φοβάμαι ότι το ίδιο ισχύει για την ετήσια εκθέσεση τη συντονισμένη άμυνα, την GARD, ε, για τον απλούστατο λόγο διότι δεν μπορούμε να εξετάζουμε ετησίως και συλλογικώ εάν έχουν επιτευχθεί στόχοι όταν δεν έχουμε καθορίσει τους λόγο στόχους. Αυτό γιατί, γιατί θέλω να πω ότι δεν τελευταία ελπίδα, τη μεγαλύτερη ελπίδα όλων των προασπιστών της Ευρωπαϊκής Άμυνας, στους οποίους ανήκω και εγώ, εδράζεται επί των όμων σας. Ο δεύτερος λόγος που με κάνει να θεωρώ ότι αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα είναι κάτι καλό και ότι προσεγγίζει την αγορά την αγορά της άμυνας, του ΣΥΠΗΝ, όχι από την πλευρά της προσφοράς όπως η οδηγία του 2009 όσον αφορά τη δημόσια προμήθεια, κατοικές προμήθειες για την άμυνα, αλλά από την πλευρά της ζήτησης. Με άλλα λόγια, θέτει χρήματα, διαθέτει χρήματα και όχι αποκλειστικά κανόνες. Και γι' αυτό ενδεχομένως, ενδεχομένως και επιμένω από αυτού, είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει το όλο παιχνίδι θα είμαι πιο σύντομο σε αυτή τη δεύτερη μου ε, παρατήρηση όσον αφορά τι συμμόρφωση με συνθήκε. Δεν ήθελα αυτή την ακρόαση να τη μετατρέψω σε μια ε, ομιλία νομικού. Ε, όμως έχω ετοιμάσει γνωμοδότηση νομικής φύσεως που σας υποβάλλω και που έχω και στην ιστοσελίδα μου και είναι στην πρόσβαση όλων και το έκανα αυτό ούτως ώστε να δείξω, να συγκρίνω σε σχέση με τους ομολόγους μου την άποψή μου όσον αφορά αυτή τη νομική θέση. Πρέπει να πιστήσω την προσοχή όμως στο εξή ότι στη δημοκρατία ο καθένας υπομίζεται τις ευθύνες του. Εκείνοι που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από νομικές γνωμοδοτήσεις, ίσως και μόνο των υπηρεσιών τους για να δράσουν ή να μην δράσουν. Θα πρέπει σίγουρα να συμβουλευτούν τις νομικές υπηρεσίες μπορούν ανάλογα με τι ανάγκε να ακούσουν και τι απόψει εμπειρογνωμόνων όπω είμαι εγώ, αλλά θα πρέπει πάνω απ' όλα να δράσουν. Να δράσουν ατρόμητα, διότι ο μόνος που μπορεί να επιβάλλει το νόμο σε ένα κάτω δικαίου είναι ο δικαστή. Αν κάποιοι από εσά έχετε αμφιβολίε όσον αφορά πώ συμμορφώνεται το πρόγραμμα με τι συνθήκε ας ε, ζητήσουν ε, να προσφύγουν στους δικαστές και το δικαστήριο θα αποφανθεί. Εγώ προσωπικά δεν έχω αμφιβολίες και έχω φέρει μαζί μου το χαρτοφυλάκι, έχω ε, τις υπόλοιπες λεπτομέρειες εδώ και μπορώ να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις νομικού περιεχομένου και έρχομαι στην τρίτη μου παρατήρηση. Θα πρέπει να επιδείξετε μεγάλη υπομονή διότι ε, δημιουργείται τα θεμέλια ενός ε, σπιτιού που θα δει το φως ε, μόνο μετά από 15 χρόνια. Θα πραγματοποιηθεί το σπίτι, θα οικοδομηθεί το σπίτι. 15 χρόνια είναι ο μέσος όρος μεταξύ της εκκινήσεως μιας δράσεως για την έρευνα στην άμυνα και τη δημιουργία του καταλήλου δυναμικού. Δηλαδή, ε, ο εξοπλισμό των δυνάμεων, ακόμα και ο σύγχρονο εξοπλισμό των δυνάμεων σήμερα, όπω κάποια πολεμικά μαχητικά αεροσκάφη, ε, είχαν ε, σχεδιαστεί πριν από 15 χρόνια το λιγότερο. Δηλαδή ότι η έρευνα που γίνεται σήμερα στα διάφορα εργαστήρια τα ερευνητικά δεν θα δημιουργήσει διαφορά στην δυναμικότητα των όπλων δυνάμεων παρά μόνο σε 15 χρόνια. Λοιπόν, είναι σημαντικότατο τα θεμέλια που θέλετε να δημιουργήσετε να είναι στέρεα και να επιτρέπουν και την ευελιξία. Από αυτή την οπτική γωνία θα πρέπει να αποφευχθούν ε, τρεις ύφαλοι και προβλήματα. Πρώτα απ' όλα να μην λάβετε υπόψη ε, τι γίνεται, τι προηγείται της αμυντικής έρευνας. Δηλαδή ο σχεδιασμός της άμυνας είναι κάτι σημαντικό. Ε, πράγματι, μία από τις ιδιαιτερότητες αυτής της έρευνας είναι ότι έχει ένα προσανατολισμό Όσον αφορά την άμυνα, δεν κάνουμε μια έρευνα σαν αυτό σκοπό, αλλά θέλουμε να παράγουμε τι αναγκαίε τεχνολογίες ε, και τις δυνατότητες που έχουν ανάγκη οι ενόπλε δυνάμεις. Άρα υπάρχει στατικικό μονοπάτι που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές αρχές μέχρι τέλους αν θέλουν είναι Όμως αυτό δεν ισχύει τελικά από τη μία πλευρά υπάρχει μια σφαιρική γενική στρατηγική και ένα επίπεδο φιλοδοξιών και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα σχέδιο δημιουργίας αναπτύξεως όσον αφορά την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Άμυνας αλλά ε, λείπει μια λευκή βίβλος μεταξύ των δύο στοιχείων. Λοιπόν, αν οι Ευρωπαίοι δεν μεταφράσουν σε στατιωτικούς όρους τους πολιτικούς στόχους που έχουν καθοριστεί, τότε δεν υπάρχει παρά μικρή δυνατότητα για την επίτευξη των στόχων. Όπω έλεγε και μεγάλο Ενέκα, δεν υπάρχει ούριο άνεμο για εκείνον που δεν ξέρει που πάει. Λοιπόν, είναι δύσκολο ο δρόμο πολιτικό, αλλά μπορεί να ακολουθηθεί. Ήδη δύο φορέ ε, μέσω των στόχων του Ελσίνκη έχει ανοίξει ο δρόμο. Αυτή είναι η απόδειξη. Και τα κάτι μέλη που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ ακολουθούν το δρόμο αυτό τακτικά στα πλαίσια ε, το NDPP, ε, τη διαδικασία λήψη αποφάσεων του ΝΑΤΟ. NATO Defense Planning Process. Εάν δεν συνδέσετε την έρευνα και ανάπτυξη την αμυντική με το σχεδιασμό της άμυνας, θα οργανώσετε ένα διαγωνισμό, διαγωνισμό ομορφιάς παραπάνω, όπως έγινε μέσω της ΠΕΣΚΟ, που τελικά, τελικά θα, θα επιτρέψει πολιτικούς να πούνε ότι κάνουν κάτι και να εισπράξουν κάποια χρήματα βιομηχανική. Γι' αυτό έχει επιφανή ρόλο να δραματίσει το κοινοβούλιο σας. Θα πρέπει να πετήσετε όχι μόνο να υπάρξει σχεδιασμός μεταξύ προγράμματο του αμυντικού σχεδιασμού και των σχεδίων αναπτύξεων δυνατοτήτων των κρατών μελών, αλλά θα πρέπει να διατηρηθείτε αυτά τα σχέδια σε τι εξυπηρετούν όσον αφορά τι ευρωπαϊκέ φιλοδοξίε. Αυτό με οδηγεί στο δεύτερο υφάλο. Να μην θεωρείτε αυτό που προηγείται, την, τι προηγείται τη Άμυνα, Ε, τι ακολουθεί μάλλον. Δηλαδή τα προγράμματα εξοπλισμών. Και αυτά είναι αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα. Το EDITP είναι το, ε, ανήκει σε ένα, είναι από τα στοιχεία της έρευνα και ανάπτυξης και θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα στοιχείο, δηλαδή τη δημιουργία δυναμικότητα. δυναμικότητας. Δεν θα επιμείνω, διότι υπάρχει διάταξη στον κανονισμό που προβλέπει ότι οι δικαιούχοι των πιστώσεων θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να αγοράσουν τα προϊόντα τους. Αυτή είναι μια έξοχη επιλογή που έλειπε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα της έρευνας όσον αφορά τον τομέα της ε, άμυνας. Τρίτος ύφαλος και τελευταίος, θα πρέπει να βρείτε σωστή ισορροπία μεταξύ τη συμμετοχή των διαφόρων βιομηχανιών όλων των κρατών μελών περίπου με την ανταγωνιστικότητα που επιβάλλει το αντίθετο, δηλαδή την επίκεντρωση των προσπαθειών στι πιο αποδοτικέ βιομηχανίε. Λοιπόν, θα είναι μεγάλο ο πειρασμό για όλα τα κράτη-μέλη. Θα θέλουν να πετύχουν κέρδη και τρόπε. Αυτή είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων. Επίση, ισχύει στην Ευρώπη όπω και στι ΗΠΑ και στη Γερουσία το λένε, όπου ευφυή, τον πιο ευφυή που γίνεται διότι αν επικαλύψετε τη βιομηχανική δυναμικότητα που ήδη υπάρχει, τότε η διόρθωση θα είναι κάτι χειρότερο από το κακό που προσπαθούμε να διορθώσουμε. Δεν μπορείτε να μειώσετε έτσι τον κατακαιρματισμό, τον τεχνολογικό και τον παραγωγικό τη βιομηχανία. Τον αυξήσετε, αν ακολουθήσετε την προσέγγιση. Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα κακό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι σε επίπεδο έρευνα θα πρέπει να επιλεγούν οι δεξιότητε ε, και όχι πολλαπλασιάζοντα ε, τι βιομηχανίε που ήδη υπάρχουν για να πετύχουμε αποτελέσματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, θα είμαι σύντομο στο συμπέρασμα. Αν η Ένωση σήμερα ανακατεύεται με την άμυνα, είναι διότι υπάρχουν κίνδυνοι και θέλουν προστασία οι πολίτε. Όμω δεν υπάρχει καμία ελπίδα η ευρωπαϊκή άμυνα να δει το φω τη ημέρα, αν τελικά να τεθεί στα κράτη-μέλη. Όπω και η ορχήστρα του Τανικού θα συνεχίζει να παίζουν τη μουσική τη κυριαρχία στα κράτη-μέλη μέχρι ότου να βυθιστεί το καράβι. Ας δούμε κατά πρόσωπο την κατάσταση. Η αμυντική έρευνα η ευρωπαϊκή δεν είναι παρά μια ισκιά αυτής που ήταν. Η τελευταία ρηξικέλευτη εφεύρεση ήταν τα, τη δεκαετία του 40 με το ραντάρ και τους τροβιλοκινητήρες για τεριωθούμενα αεροπλάνα. Δηλαδή τώρα υπάρχει μια ευκαιρία να τη σώσετε, αρπάξτε την ευκαιρία. Αυτό αφορά την αυτονομία μας, την εξαρτησία μας και αυτό ισχύει για την ελευθερία μας. Αυτό αφορά την επιβίωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Διότι η Ευρώπη δεν ε, προσπίσει του ε, πολίτε τη, οι πολίτε τότε διερωτηθούν σε τι μα εξυπηρετεί τελικά η Ευρώπη, σε τι σημαίνει η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you for your speech. Σας ευχαριστώ πολύ για τον... την ομιλία σας, παρατηρήσεις σας και περνάμε τώρα στη δεύτερη ομιλία. Ο Μπεν Ε, λυπούμε για το ότι Ιανουάριο 2018 κάθομαι σε ένα αρσενικό πάνελ. Και βεβαίω ε, τίθεται και το ζήτημα της λήψης αποφάσεων σε αυτόν τον ε, τομέα. Εμείς είμαστε κατά του μιλή στο πρόγραμμα αυτό έρευνας ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσφέρει κάποια σοβαρά μαθήματα τα οποία ίσως δεν ελήφθησαν υπόψη στις ε, τρέχουσες ε, διαβουλεύσεις. Επίσης ε, θα ήθελα να πω κάποια γενικά πράγματα για την πολιτική συγκυρία την οποία νομίζω ότι εκμεταλλεύεται κοινικά η αμυντική βιομηχανία. Είμαι βεβαίως υπέρμαχο του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδράσει συμβολικά, πρακτικά, στο Brexit, στον Τραμπ, το ΝΑΤΟ το οποίο σιγά σιγά αποσυντήθεται, αλλά είμαι πεπισμένος ότι η βιομηχανική αυτή στρατηγική δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε μια καλύτερη αμυντική πολιτική, περισσότερη ασφάλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες και θα επανέλθω να σας πω γιατί. Θα κάποιος ο οποίος έχω παρακολουθήσει από κοντά το πώς ε, έχουν ε, θολώσει γραμμές μεταξύ άμυνας και ασφάλειας, ε, πολέμου και ειρήνης ειλικρινά φοβάμαι από την τυφλή πίστη που εξακολουθεί να δείχνει η Ευρωπαϊκή είναι εκπληκτικό το ότι σε λιγότερο από ένα έτος έχουμε προχωρήσει τόσο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και αντιλαμβάνομαι και την πίεση την οποία υφίσταστε σε σχέση με το ΠΔΠ, το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι λυπηρό τουλάχιστον το ότι οι προπαρασκευαστικές δράσεις ήδη ε, έχουν ξεκινήσει γιατί αυτό το οποίο σημαίνει ε, είναι ότι θα δώσουμε όπλα σε κάποια από τα πιο στιγνά καθεστώτα του πλανήτη. Το 2018 τα κράτη-μέλη της Ένωσης ε, έστειλαν 82 δισεκατομμύρια ευρώ στην περιοχή Μέσης Ανατολής. Είναι εκπληκτικό το ότι εξετάζεται αυτές τις πολιτικές χωρίς ταυτόχρονα να εξετάζεται την ενίσχυση του κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων που προφανώς δεν λειτουργεί ήδη ανέφερε και ο Στανεφός του πράσινου, ότι θα γίνει με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα και επίσης στην στρατηγική αυτονομία αλλά τις ξέρετε αυτές τις ε, συζητήσει και μάλλον έχετε ήδη καταλήξει τα συμπεράσματά σας για το πώς ε, θα έχετε μία θέση υπέρ της άμυνας ή κατά του μιλιταρισμού. Και στο χρόνο που μου απομένει θα ήθελα να δω πριν από 12 χρόνια σε αυτό εδώ το κτίριο και ε, πραγματικά είχα λυπηθεί για το ότι δημιουργήθηκε μια ομάδα η οποία δεν λογοδοτούσε πουθενά και θα ξεκινούσε μια προκατακτική έρευνα και αμφισβήτησα τις βασικές υποθέσεις αυτού του προγράμματος. Ακριβώ για να υπάρξει δημοκρατικός έλεγχος και να δούμε το τι αντίκτυπο θα έχει στην ε, κοινωνία. Είχα προεδρεύσει σε ομάδες διοντολογίες, έχω αξιολογήσει προτάσεις έργων, έχω εκπαιδεύσει αξιωματούχους ε, της Κομισιόν για τα, όπλα διπλής, ε, τα προϊόντα διπλής χρήσης πλαίσιο 9. Σας τα λέω αυτά γιατί θέλω να αντιληφθείτε ότι κάνω επικοδομητική κριτική της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα αυτών. Ας το πώς πέρασε μέσα από το Κοινοβούλιο σε μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια. Ας θυμηθούμε τα τότε επιχειρήματα. Τι μας έλεγαν. Μας έλεγαν ότι πρέπει να επιδοτήσουμε τον αμυντικό κλάδο για να μην εξαρτώμεθα από Κίνα και ΙΠΑ. Μας είπαν ότι πρέπει να αυξήσουμε σχετική αγορά. Μας έλεγαν ότι η αστυνομία και οι ένοπλες ε, δυνάμεις δεν είχαν τα απαραίτητα μέσα. Μας έλεγαν ότι θα έπρεπε να επιδοτήσουμε τη μεταφορά στρατιωτικής τεχνολογίας ε, στον πολιτικό τομέα ασφαλείας ε, για να μας προστατεύσει από την τρομοκρατία και την Και βεβαίως μας υποσχέθηκαν την αριστεία και την καινοτομία την οποία αναφέρατε κι εσείς. Όλα αυτά λοιπόν κάπου τα έχω ξανακούσει. Και Έχοντας αυτά κατά νου, αναρωτιέμαι εάν μπορεί κάποιος σε αυτή την αίθουσα να μου πει μία καινο... παράδειγμα καινοτομία που προέκυψε από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι μέχρι στιγμής. Ε, δεν ξέρω, ίσως οι συναδελφοί μου μπορούν να απαντήσουν εδώ. Αλλά νομίζω ότι μιλάει από μόνο του το ότι δεν μπορούμε να αναπτύξουμε το πρόγραμμα αυτό βασιζόμενοι ε, λίγα ακόμα λόγια θα πω και ευχαριστώ να δεχτώ ερωτήσεις. Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το πρόγραμμα αυτό το 2004, Ανισχούσα πολύ για το τι σημαίνει αυτό για τις αστικές ελευθερίες. Η στρατιωτικοποίηση της ασφάλειας. Τώρα ανισχώ περισσότερο για κάτι άλλο. Ότι η όλη αυτή υπόθεση μάλλον είναι μια τεράστια σπατάλη χρημάτων. 3 δισεκατομμύρια ευρώ των φορολογουμένων. Οπότε αντιλαμβάνομαι αυτά τα οποία είπε ο Ευρωβουλευτή που με εκπροσωπεί στο ΕΕ, αν και έφυγε την αίθουσα. Κάντε μια βόλτα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα, όπω κάνω εγώ. Η τύχη είναι, δεν είναι στους γιατί δεν υπάρχουν. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι γιατί είχαμε αυτήν την τεράστια σπατάλη χρημάτων και στην ε, αμυντική βιομηχανία ουσιαστικά να καθορίσει το πρόγραμμα. Χρησιμοποίησαν τα κονδύλια ως μια γενική ε, επιδότηση για πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως θα έκαναν. Και έτσι εκπλήσωμαι για το ότι δεν έχει συζητηθεί περισσότερο ποιε ήταν οι, οι ερευνητικές προτεραιότητες για το πρόγραμμα αυτό. Δεύτερον, κατάφορη έλλειψη δημοκρατικής λογοδοσίας. Δεν καθόρισε τις προτεραιότητες στο Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει μηχανισμός αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, των παραδοτέων. Υπήρχε καινοτομία, υπάρχει κάποια αξία σε αυτές τις δαπάνες. Έχουμε κάποιες μεσοπρόσμες αναθεωρήσεις, άχρωμες, άοσμες, που δεν μας λένε τίποτα. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Ή το τι έγινε με αυτά τα λεφτά, τι έχουν πετύχει πέρα από καθαρά στατιστικά αποτελέσματα. Ρωτήστε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αστυνομική Τεχνολογία που συστάθηκε ακριβώς λόγω αυτών των αποτυχιών. Δεν υπήρχαν αποτελέσματα γιατί τα έργα πήγαιναν, είχαν προσανατολιστεί στις ανάγκες της βιομηχανίας και όχι του κλάδου. Εδώ πέρα λοιπόν βάζουμε το κάρο πριν από το άλογο. Κάνουμε τα πράγματα ανάποδα. Ακόμα και αν υποστηρίζετε λοιπόν επί της αρχής αυτήν την πολιτική όπως ε, αντιλαμβάνουμε ότι πολύ κάνετε, θεωρώ ότι πρέπει να την απορρίψετε γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διακριτική ευχέρεια που δίνεται στην βιομηχανία να καθορίσει το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει μηχανισμός δημοκρατικής εποπτείας που χρειάζεται ένα τέτοιο πρόγραμμα και μοιραία και αναπόφευκτα θα καταλήξει σε σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων. Εάν στηρίζετε την αμυντική συνεργασία, θα ήθελα να ζητήσετε από την Κομισιόν να ξαναρχίσει από την αρχή και να κάνει μια αξιολόγηση αναγκών και να πάει πέρα από το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Και αν μπορεί να δικαιολογήσει κάτι, τότε να δώσετε τα λεφτά. Τελείωσε ο χρόνος μου. Θα πω το εξής. Απλά πετάτε τα χρήματα σε ένα κουβά και λέτε κάντε κάτι εκεί πέρα. Δεν βοηθάει αυτό την ευρωπαϊκή άμυνα, ούτε τον ευρωπαίο φορολογούμενο και δεν θα έχει αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να σταματήσω την ε, κριτική σας. Μακρηγορήσετε περισσότερο από τους υπολοιπούς, αλλά σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Είναι εξαιρετικές ε, η σοβαρή συζήτηση όχι μόνο στην ε, Επιτροπή μας εδώ, αλλά και στη συνέχεια θα συζητήσουμε και με των τροπολογιών και τα λοιπά και θα λάβουμε υπόψη τις πολύ σοβαρές παρατηρήσεις σας. Και αναφερθείτε και στο πρόβλημα της ισότητας των δύο φέλων. Θα ήθελα να πάρετε πρώτη το λόγο, γιατί είναι και πολύ σημαντικό αυτό το τμήμα της συζήτησης. Κύριε Πρόεδρε, εδώ είμαι ιδιαίτερα ταπεινή γιατί πρόκειται για μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση και πιστεύω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής μας θα έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, όσο και εγώ. Ευχαριστώ τους δύο μιλητές, τον κύριο Μάουρο και τον κύριο Χάις. Θα θέσω την ερώτησή μου, αλλά θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για την παρέμβαση του τελευταίου μιλητή. Έχουμε και το κεφάλαιο αυτό της συνθήκης το οποίο ενεργοποιήθηκε έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι δεδομένου του πώς άλλαξε. Να πω νομίζω άλλο, ο κ. Πούτιν ξεκίνησε τις επιθετικές ενέργειες ε, το 2010. Σας ευχαριστώ κ. Σκολίτσικ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω στον συνάδελφο από τη Γερμανία πως ε, αν ε, κάνει τους ορθούς ε, υπολογισμούς θα φτάσει στην ακόλουθο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει περισσότερα χρήματα για την άμυνα από ότι ο Πούτιν και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πανούν πάνω από το ίμιση των συνολικών δαπανών ε, όλου του πλανήτη. Λοιπόν, τώρα έχει δίκιο ο κ. που είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα να έχει ένα πρόγραμμα σε αυτόν τον τομέα, αλλά ο κύριος ε, Χαές επίσης έχει δίκιο. Είπε ότι όταν έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι δυνατόν να ελέγχεται και θα πρέπει να μπορούμε να αξιολογούμε και τα αποτελέσματα. Ανεξάρτητα με το αν υπήρξε πιλωτικό πρόγραμμα ή όχι. Και εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία του τι θα έπρεπε να έχουμε στο έγγραφο. Αναφέρθηκε σε αυτό και ο κύριος Πάσκου, γιατί αν ε, μιλάμε για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει σαφείς στόχους και θα πρέπει να είναι σαφές το πώς θα παρακολουθούνται και θα υποπτεύονται οι στόχοι αυτοί. Είπε ο κύριος Λαντόφσκι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς όπου τα κράτη-μέλη μπορούν ε, να έχουν μία ενιαία προσέγγιση. Μπορούμε να μιλάμε για τομείς όπως η αεροπλοεία, ή τα διαστημικά προγράμματα. Από την άλλη όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε μεγαλύτερο κράτος μέλος αναπτύσσει και κάνει έρευνα για τα δικά του πυρομαχικά, κάνει έρευνα και αναπτύσσει δρόν και άλλα Και αν κάποιες από αυτές τις προσπάθειες ήταν συντονισμένες και αν κάποια από τα μέρη που έχουν εισαχθεί μέχρι τώρα μπορούσαν να αντικατασταθούν από μέρη και που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το πρόγραμμα θα είχε καλά αποτελέσματα και θα είχε προσθεμένη αξία. Και συμφωνώ με τον κύριο Χάιες ότι για την ε, ασφάλεια των πολιτών μας, το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλές διεθνείς συμφωνίες και να μπορούμε να καταπολεμήσουμε και να προλάβουμε την τρομοκρατία, όχι με τα όπλα, αλλά με άλλα εργαλεία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Ε, θέλω να πω στου προσκεκλημένου ότι ε, ο κύριο προσωπεί τον εαυτό του. Εγώ λυπάμαι που αποφάσισαν οι Βρετανοί να μα εγκαταλείψουν, ε, αλλά υπόθηκαν. Ε, το άρθρο 14 λέει το πρόγραμμα ότι πρέπει να επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Έχουμε λοιπόν και τέτοιες ανησυχίες ε, και εδώ επανέρχομαι στις προτάσεις του κυρίου Μάουρο με τις οποίες συμφωνώ. Εμείς οι πολιτικοί πρέπει να θέσουμε τους στόχους ε, και φυσικά τα προγράμματα, η βιομηχανία της άμυνας που είναι αρμόδια να θέσει τους στόχους. Συμφωνώ μαζί σας λοιπόν σε αυτό. αν παρακαλούσατε τους κυρίους εμπειρογνώμονες να μας δώσουν τις σημειώσεις τους, διότι θα ήθελα να ρίξω ξανά μια μακροδότηση από τον Δημόσιο Κορβανά, ότι πρέπει να είμαστε ιδιοκτήτες των πνευματικών δικαιωμάτων και δεν θέλουμε άλλα όρια, δημόσια χρήματα 100% και η βιομηχανία είναι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων. Από πλευράς ανταγωνισμού θα υποστηρίζετε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, να συμμετέχει στο ε, Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού ε, Αμυντικού Ταμείου. Δεν είδαμε κάποια πρόταση, κάποια διάταξη που να δίνει στα ερετά μέλη χρηματοδοτούμενη από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Είμαι περίεργος. Πού ακριβώς θέλει να δαπανίσει τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και απηχώ και το και πολλές δεκαετίες όποτε κάποιος ήταν υπερβολικά κριτικός, κάποιος από το κόμμα σας θα έλεγε πηγαίνετε στην Ανατολή. Ο κ. Αλέξης, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζωή συζήτηση συνθισμένη στην Επιτροπή μας από την Γενική Διεύθυνση Ανα... Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι ομιλητέ σας απαντήσουν. Ο κύριος Μάωρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις ξεκινώντας από τις ερωτήσεις που μετέθησαν από τον συνάδελφο, τον κύριο Χαΐς, που τον ευχαριστώ και θέλω να σωστά θέτει το θέμα της αποτυχίας του προγράμματος για την έρευνα στον αμυντικό τομέα. Θα πρέπει να μαθαίνουμε από τα σφάλματά μας. Όταν έπρεπε συντάξω μια έκθεση για το κοινοβούλιο σας το 2016 για το μέλλον της αμυντικής της έρευνας στον αμυντικό τομέα, πήγα να συναντήσω του υπευθύνους τα κράτη-μέλη, διότι τα κράτη-μέλη δεν ήταν στο κύκλωμα. Και έτσι απαντώ κατά κάποιο τρόπο στην ερώτηση τη κυρία Ιγήτριας. Ο λόγο για τον οποίο τα ερευνητικά προγράμματα του τομέα τη ασφαλεία ήταν αποτυχημένα είναι ότι αυτή η έρευνα δεν είχε προσανατολισμό και ακριβώ αυτό ήθελα να στείλω. Χανία ε, είναι κάτι διαφορετικό. Όπως ε, είναι διαφορετικά θλήματα, όπως είναι το ράγμπι με το ποδόσφαιρο. Αν κάνετε αμυντική έρευνα με στόχο να δημιουργείτε θέσει απασχόληση, με στόχο ε, να βγάλετε ψωμί, το, για τους άλλους μην το κάνετε. Διότι θα επιδεινώσετε τα προβλήματα των σχεδίων δημιουργίας δυναμικότητας αν θέλετε να παίξετε ένα ρόλο. Θα πρέπει, αυτός ο ρόλος είναι να υποχρεώσετε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όλος ιδιαίτερος ε, το, το κέντρο έρευνας να συντάξουν ε, μία λευκή βίβλο, να μεταφράσουν σε στατιωτικούς στόχους ε, τους πολιτικούς στόχους, τι είδους ε, επιχειρήσεις θέλετε ε, παρυφές από τη Ρωσία, πώς θα προστατευτείτε την τρομοκρατία εντός των συνόρων μας. Πρέπει να έχετε στόχους. τώρα, τώρα, που διαφωνώ ή συμφωνώ λιγότερο. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το ρόλο του Κοινοβουλίου και των κρατών κυβερνήσεων και δεύτερον όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, όσον αφορά το ρόλο των κοινοβουλίων και λίγα των βουλευτών. Και είχε ηγηθεί ο κύριο Γκάλερ για να δοθούν χρήματα στο ειδικό τομέα. Τα κράτη-μέλη δεν θέλουν. Είναι πολύ δυσταθερά τα κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να λέμε λοιπόν το κάνουμε αυτό διότι ικανοποιεί τα κράτη-μέλη. Όχι. Τα κράτη-μέλη πάνω απ' όλα δεν θέλουν η Ένωση να αναμειχθεί στον τομέα τη άμυνα. Θέλουν αυτοί μόνο να πω ότι αυτή η ιδέα είναι γελία που αναφέρθηκε, δηλαδή ότι αγοράζουμε ή παράγουμε εξοπλισμό αμυντικό ε, όπως αγοράζουμε σαπούνια ή αυτοκίνητα πολυτελείας. Δεν θα αγοράσει κανείς ένα πυρηνικό υποβρύχιο ή μη πυρηνικό όπως αγοράζει κανείς μια Jaguar. Αληθεύει ότι πούμε κάποιες ε, κάλτσες για το στρατιώτη ή κάποια κράνη και, όχι, ε, και φορτηγά και όχι άρματα μάχης. Κατά λοιπά όμως είναι μια ιδιαίτερη βιομηχανία που έχει λόγο ύπαρξη διότι το απαιτεί το κράτο. Δεν θα κατασκευάζουμε μαχητικά αεροσκάφη για να τα εξάγουμε. Ε, το υποστηρίζετε. Εάν αγοράζετε όπλα από μία χώρα, τότε εξαρτάστε από αυτή τη χώρα. Οπότε ερχόμαι στο τρίτο μου θέμα, η ρόλη του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Συγητρία δύσκολο να καθοριστεί, διότι υπάρχουν δύο πρωτοβουλίε που ανταγωνίζονται μία την άλλη. Και μετά το Ευρωπαϊκό αυτό το Ταμείο τη Άμυνα που ξεκινήσατε, ποιο είναι ο ρόλο αυτών των δύο πρωτοβουλειών και η σχέση τη μία με την άλλη που επηρεάζει του ρόλου των θεσμικών οργάνων. Είναι πλειοψηφία. Και αν δεν το κάνετε αυτό, τα κράτη-μέλη θα το κάνουν. Θα κάνουν αυτό που έκαναν και στην εκκίνηση του ΠΕΣΚΟ. Όσον αφορά τα 40 προγράμματα τη ΠΕΣΚΟ, τα αρχή να διαλέξει τι έχει ανάγκη. Δεν υπήρχε γενικό συμφέρον και ενδιαφέρον ευρωπαϊκό. Αυτό που ενδιέφερε ήταν το Σέγγεν τη άμυνα στα κατημέλη. Τα υπόλοιπα αφορούσαν το ΝΑΤΟ, τα προγράμματα. Και όχι το PSTC, το ΠΕΣΚΟ. Κύριε Κόντιτσεκ, ποιο είναι ο σκοπό του προγράμματο, η επιτροπής. Επιτροπή. Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει μέσω τροπολογιών να ενισχύσετε το κείμενο. Ευπρόσδεκτε οι τροπολογίε, όπω θα κάνει και το Συμβούλιο. Πάρα πολύ καλό. Στατηγική αυτονομία. Τι είναι η στατηγική αυτονομία. Απλούστατα για να καταλάβει ο καθένας με εύληπτους όρους η δυνατότητα να κάνει κανείς πόλεμο μόνος. Μια συνιστόσα πολιτική, η δυνατότητα λήψεως αποφάσεων είναι αυτή και εκτελέσεως των αποφάσεων. Δεύτερον, μια συνιστόσα επιχειρησιακή που είναι προφανής να διαθέτει κανείς δυνάμεις ανάλογα με την αποστολή που έχει καθοριστεί και τρίτον, μια συνιστόσα βιομηχανική. Υπάρχει βιομηχανική. Αυτά. Πού να επενδυθούν τα χρήματα πρέπει να επενδύονται εκεί που υπάρχει μέγιστη μόχλευση. Έκανα προπαρασκευαστική μελέτη για λογαριασμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν, δεν είναι δημόσια όσον αφορά του τομεί όπου θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσει. Εκεί που θα έχετε περισσότερη μόχλευση είναι με προγράμματα που συνδέουν. Έχουν σημαντικό κόστος μάλλον, αλλά συνδυάζουν πηλίκων ε, ε, κόστος έρευνας και ανάπτυξης ε, με παρονομαστή το συνολικό κόστος της έρευνας πολύ ψηλό, όπως οι δορυφόροι. Ενσωτικός δορυφόρος, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης Ποιε είναι οι επιτυχίε, ποιο μπορεί να μου απαντήσει αυτό το ερώτημα, γιατί τώρα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα χωρί να ξέρουμε πού πάνε αυτά τα χρήματα, πού είναι η χούσε η αμυντική βιομηχανία και διάφορα Ινστιτούτα έρευνε που υποστηρίζουν ε, την αμυντική βιομηχανία και είχαμε λιερχείται από στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας, κάνει στη συνέχεια συστάσεις ε, για το ποιες ε, προτεραιότητε έρευνα θα πρέπει να επειδή του παρελθόντος. Βλέπω όμω ότι ακριβώς τα ίδια λάθη γίνονται στο σχεδιασμό αυτού του προγράμματος. Και κάτι τελευταίο. Θα πρέπει να... Ε, μπορεί παραδείγματο χάρη ε, να βασιστεί και πείτε να εδώ είναι το κενό και να και η ξεκάθαρη λύση μπορείτε να πείτε ξεκάθαρα αυτές είναι οι πρινάς, όμως αυτό φαίνεται ότι δεν λειτουργεί. Θα σταματήσω εδώ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Α, ξεκινήσουμε από τις ευχαριστίες προς την συγγήτρια. Ήταν πολύ ξεκάθαρη και έφυξε όλα τα σημεία εξαντλητικά. Λοιπόν, ξεκινάμε από το σκεπτικό ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό λειτουργεί. Πρόκειται για μια οδηγία η οποία, τα σημεία που έθιξε η συγκήτρια πολύ σύντομα, είναι σωστή η έμφαση στην πρώτη παράγραφο για την αναγκαιότητα να διατηρήσουμε ε, τους καταναλωτές στο επίκεντρο των εγγύσεων που γίνονται από τον οικολογικό σχεδιασμό Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το φορούν τις τεράστιες επενδύσεις που πρέπει να συνεχίζουν να αποφασίσουν να κάνουν επιχειρήσεις προκειμένου τα προϊόντα να σέβονται αυτά τα κριτήρια τα οποία σήμερα συζητούμε. Τώρα το σημείο που αφορά την ορθή εισαγωγή κριτηρίων που αναφέρει σήμερα συζητούμε. Τώρα το σημείο που αφορά την ορθή εισαγωγή κριτηρίων που αναφέρεται ε, της, της απόδοσης του προϊόντος και της τιμής του. Αυτά όμως είναι κριτήρια που έχουν έναν ορισμό πολύπλοκο και είναι... Δεν ισχύει το ίδιο με τα δύο ε, διασπόμενα. Και ο νόμος ο είναι πάρα πολύ καλό Το ερώτημα είναι αν πρέπει και άλλες χώρες ε, να το ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο κύριος Κόλτσεκ ε, έχει δίκιο. Εάν δεν απαχωρεύσουμε τα διάφορα είδη πλαστικού δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα ανακυκλώσουμε. Έχω τρεις ερωτήσεις ε, προς την ε, Κομισιόν και σας ευχαριστώ Μισελ για την έκθεσή σας. Τα λευκά είδη. Ο Λόνας Μπερκλέης της είπα μου είχε πει ότι το Dieselgate ε, για τα αυτοκίνητα θα συμβεί μάλλον και στις ε, συσκευές γιατί όταν έχουμε ένα συνδεδεμένο ψυγείο έχουμε έναν υπολογιστή μέσα στο ψυγείο και μπορούμε να δώσουμε οδηγίες βεβαίως για το τεστ στο τσιπάκι αυτό. Συμφωνείτε λοιπόν με τον άνθρωπο ότι τα συνδεδεμένα, οι συνδεδεμένες συσκευές ε, είναι πιθανότερο να κλέψουν στο τεστ. Δεύτερον, για μένα ο οικολογικός σχεδιασμός είναι περισσότερο μια στρατηγική εξαγωγών για την Ευρώπη. Τι κάνει η Κομισιόν έτσι ώστε άλλες περιοχές ε, του πλανήτη να, εγκρι... να υιοθετήσουν αυτές τις προδιαγραφές για να έχουμε και ένα πλέον έκτημα εμείς. Και τέλος, κατά την άποψη της Κομισιόν, πότε σκοπεύετε ακριβώς να ξαναδείτε την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού. Σε αυτή την θητεία ή σκοπεύετε για μετά το 2019, ε, μετά τις ευρωεκλογές. πρώτη Κοιτάξτε, σχόλια θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Χότσον, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενική Διεύθυνση Υπευθυγενών.